12. Κυρίες και κύριοι, η προσεχή συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο, 13 ε, Δεκεμβρίου, από τις 9 ως τις 2 και από τις 3 ως τις 8 και στη συνέχεια από τις 9 ως τις 12 το βράδυ. Η εμερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας και σας εύχομαι καλή νύχτα.